ΔΕΠΡΕ προβλέψεις σε σώμα και δαπανών για το οικονομικό του 2016 τμήμα 1 κοινοβούλιο πρώτος έχει τον λόγο για 4 λεπτά ο εισηγητής ο κ. ΔΕΠΡΕ έχετε τον λόγο ε, Κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι ο, οι υπολογισμοί εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το 2016 ένα αντικείμενο από την Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασης και διαπιστώσαμε ότι θέλαμε να προτείνουμε ένα προσχέδιο προϋπολογισμού ρεαλιστικό με ένα αλλά πολύ αυστηρό προς τις αυξήσεις των κοντιλίων. Γι' αυτό από την αρχή είχαμε συμφωνήσει πρώτον ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2016 πρέπει να βασίζεται στο 20% του συνόλου των διοικητικών εξόδων της Ένωσης. Δεύτερον, ότι η αύξηση των τρεχών των κονδυλίων λειτουργίας σε σύγκριση με το 2015 δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1,6% αλλά προσθέτουμε ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών μας αναγκάζουν να προσέξουμε ιδιαίτερα και το πρόβλημα της ασφάλειας και γι' αυτό πέρα από το 1,6% αύξηση του τρέχοντος προπολογισμού αποφασίσαμε να δημιουργηθεί ένα μια ειδική θέση 15 εκατομμυρίων ευρώ για να ενδυναμώσουμε ιδιαίτερα στις Βρυξέλλες την ασφάλεια των κτηρίων του Κοινοβουλίου και να δοθεί και σημαντικό τμήμα των κοντιλίων αυτών στην ηλεκτρονική ασφάλεια στην κυβερνοασφάλεια μεταξύ άλλων και των χώρων του Κοινοβουλίου. Αυτό το θεωρήσαμε απαραίτητο. Μετά από αυτό το γενικό πλαίσιο επικεντρωθήκαμε στις λειτουργικές προτεραιότητες που θέλαμε για το 2016 και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να ενισχυθεί μία προτεραιότητα, δηλαδή η ενίσχυση των κονδυλίων για την, ε, που θα μας επιτρέψουν να ασκήσουμε τα κοινοβουλευτικά μας καθήκοντα διότι όπως ξέρετε από τη Λισαβόνα και μετά έχουμε περισσότερες δικαιοδοσίες και άρα και περισσότερες ανάγκες προσωπικού και όμως δεν έχουμε αρκετά μέσα για να ελέγξουμε όπως θα έπρεπε τις κατεξουσιοδότησης πράξεις και τις νομοθετικές πράξεις. Εξού και πολλαπλά μέτρα που προτείνουμε και συμφωνούμε με το Συμβούλιο επ' αυτόν. Πρώτον, η ενίσχυση κατά 20% της θέσης του κοινοβουλευτικού γραμματέα που θα ελέγχει ακριβώς ε, τα κατεξουσιοδότηση πράξεις κλπ. Δεύτερον, ζητήσαμε από το περιθώριο και δέχτηκε να εφαρμοστεί ένας νέος κανονισμός για καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ των τοπικών και των μη τοπικών βοηθών. Όλοι καταλαβαίνουν ότι η κανονική βοηθή είναι απαραίτητη για κάθε βουλευτή για να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ως συνομοθέτου και ελέγχου του εκτελεστικού. Τρίτον, παράλληλα με αυτά που είπα, Επίσης αποφασίστηκε τη αιτήση ορισμένων πολιτικών ομάδων και τελικά και του Προεδρείου να αυξηθεί η... το ποσό που χορηγούμε για τη γραμματεία του κάθε βουλευτού, την αποζημίωση γραμματείας. Ορισμένοι συνάδελφοι βέβαια αυτό το θεω... δεν το θεώρησαν καθόλου απαραίτητο. Άλλοι αντίθετα τάχθηκαν υπέρ του λέγοντας ότι η αποζημίωση αυτή δεν έχει προσαρμοστεί από το 11 ενώ οι μισθοί των συνεργατών μας έχουν και επίσης ζητήθηκε αύξηση του αριθμού των κανονικών βοηθών. Μεταξύ προεδρίου και Κομπού έγινε μια συμφωνία η οποία βασίζεται στο εξής. Τα απαραίτητα ποσά για τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης του προλογισμού θα απελευθερωθούν μόνον αφού εγκριθεί μία διευθέτηση με το Προεδρείο για τον αριθμό των κανονικών βοηθών έτσι ώστε να μπορούν να διευθυνθούν και τα προβλήματα των τοπικών βοηθών. Και τέταρτο και τελευταίο μέτρο κύριε Πρόεδρε, η εκτίμηση της αξίας της εργασίας ενός βουλευτού δεν είναι μόνο θέμα ποσοτικό αλλά και ποιοτικό δηλαδή περιεχομένου και το τωρινό σύστημα ranking των βουλευτών δεν ε, είναι το καλύτερο δυνατόν. Γι' αυτό το Προεδρείο και η Επιτροπή Προπολογισμών συμφώνησαν να ζητήσουν από τη διάσκεψη των Προέδρων να προσεχθεί η εφαρμογή ενός νέου κανόνα που να σταματάει πλέον να μειωθεί, να μειωθεί ο αριθμός των γραπτών ερωτήσεων Μεταξύ των προτεραιοτήτων που σας ανέφερα, το Προεδρείο και η Επιτροπή Προπολογισμών τελικά συμφώνησαν να μειωθεί από 11, ε, κατά 11.000 ευρώ ότι θα καταλήξουμε σε μείωση 11.000 ευρώ με τα μέτρα αυτά. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και των άλλων πολιτικών ομάδων καθώς και το προσωπικό της Γραμματείας της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τους συνεργάτες μας από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσίασή σας. Θα ακούσουμε τώρα τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ρούμπικ, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντεπρέ. Διαπραγματευτήκαμε πολλές ώρες και δίκαια και νομίζω πως ε, το αποτέλεσμα το δείχνει αυτό. Βεβαίω. Νομίζω πως ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να ε, εργαστούμε για να αποδώσουμε και εμείς σωστά και βλέπουμε πως Κάθε έτος μειώνονται οι θέσεις του προσωπικού κατά 1%, ο προϋπολογισμός κατά 7%, οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δίνει ένα 6% για διοικητικές δαπάνες. Από αυτό το 6% το Κοινοβούλιο παίρνει το πολύ 20% και μάλιστα είμαστε κάτω από αυτό το ποσοστό και θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ πέρα τον εισηγητή γιατί δεδομένης της γενικής κατάστασης απαιτείται και εμείς να κάνουμε η οικονομία. Τώρα, για το κονδύλιο της γραμματείας συζητάμε πάντα το πλαφόν και χαιρετίζω το ότι οι διάφορες ομάδες εδώ πέρα έχουν διαφορετικές απόψεις. Εμείς θεωρούμε πως θα πρέπει να αποφασίζει ο κάθε βουλευτής ε, μόνος του, οποίος χρειάζεται λιγότερους βουλευτές, λιγότερους ασκούμενους, λιγότερες υπηρεσίες, μπορεί να το κάνει και να λαμβάνει ένα μίνιμουμ. Από την άλλη βεβαίως υπάρχουν κάποιοι λίγοι βουλευτές εδώ πέρα οι οποίοι έχουν τεράστιο ε, βάρος ε, εργασίας και χρειάζονται τους ε, παραπάνω βοηθούς. Γι' αυτό θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν ε, το πλαφόν. Επίσης, βλέπουμε πως ε, οι υπηρεσίες της διοίκησης δίνονται αν τις ζητήσει κανείς. θα πρέπει να υπάρχει και το θέμα της διαφάνειας αλλά και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ο κάθε βουλευτής βεβαίω να τα κάνει μόνος του και να μην στέλνει τη δουλειά του στην διοίκηση. Σας ευχαριστώ για τους Σοσιαλδημοκράτε, Βλαντιμίρ Βαμάνκα για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από κοινού έχουμε σαν στόχο την βελτίωση της ζωής των πολιτών μας. Μερικές φορές όμως για την προσπάθειά μας αυτή δεν διευκολύνουμε τον εαυτό μας. Σαν παράδειγμα, οι γραπτές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι πάρα πολλές, έχουν φτάσει τις 1700 το μήνα. Αυτό φυσικά αφορά ε, πάρα πολύ κόσμο και κοστίζει κιόλας. Για να διεκπεραιώνεται η διαδικασία απαιτείται πάρα πολύς ε, κόσμος και οι απαντήσεις τις οποίες παίρνουμε πολλές φορές δεν είναι αυτές οι οποίες αναμένονται. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν, απαντούν με πάρα πολύ, δεν απαντά με πάρα πολύ μεγάλη ειλικρίνεια ή απαντά θα έλεγα χωρίς ε, ιδιαίτερη φροντίδα. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε κάποιες ε, λύσεις. Και θα πρέπει επίσης και οι οι ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γίνουν πιο ε, δημοφιλείς, να χρησιμοποιηθούν σωστά, να ξεπεράσουμε μέσω της πληροφορικής ε, τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να εξοικονομήσουμε χρήματα και το προσωπικό των επιτροπών να ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα. Η λύση στην οποία καταλήγουμε είναι μια συμβιβαστική λύση ε, Εάν πράγματι θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε, ε, ας να αλλάξουν τα πράγματα, ας υπερψηφίσουμε την πρόταση της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό τώρα για τους Ευρωπαίους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κ. Βίστησεν. Θα ήθελα να, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει. Νομίζω πως ε, το καλύτερο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι πως αντιστάθηκε σε κάποιες από τις πιο εξωφρενικές απαιτήσεις για αύξηση του προϋπολογισμού. Θεωρούμε πως οι απραγματεύσεις μεταξύ του προεδρίου και της Επιτροπής Προπολογισμού με τον κύριο Ντεπρέ ήταν ε, καλές και πραγματικά θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα. Παρά το ότι δεν μπορούμε βεβαίως να υπερψηφίσουμε τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου γιατί έρχεται σε μια στιγμή στην οποία έχουμε κρίση στην Ευρώπη και κάθε κράτος μέλος αναγκάζεται να περικόψει ε, και θεωρούμε πως είναι απαράδεκτο να αυξάνουμε τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου παρά το ότι όπως είπα τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει αύξηση στο επίδομα γραμματείας για πρόσληψη νέου βοηθού. Εμείς θεωρούμε πως είναι λάθος μήνυμα και δεν μπορούμε άρα να στηρίξουμε αυτό το συμβιβασμό. Σας ευχαριστώ. Για την αριστερά, τώρα για 1,5 λεπτό, ο Γιουνούς ο Μαρτζή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την ποιότητα της παρουσίασής του. Θα ήθελα να τον συγχαρώ γιατί η προσπάθεια την οποία είχε να κάνει δεν ήταν πάρα πολύ εύκολη. Έπρεπε να εξοικονομήσουμε 10 εκατομμύρια σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις του Προεδρείου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν, γιατί είδαμε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων να διαμορφώνονται κάποιες θα έλεγα μη αναμενόμενες συμμαχίες οι οποίες επέτρεψαν στην αύξηση κάποιων ποσών που δεν είναι και ιδιαίτερα κατάλληλες οι αυξήσεις αυτές και που σε καμία περίπτωση δεν ήταν αντικείμενο συμβιβασμού μεταξύ μας. Αναφέρομαι στην αύξηση της αποζημίωσης για τη γραμματεία, την αύξηση κατά αρκετά εκατομμύρια για την ανακαίνιση των επίπλων, όπως επίσης και η χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων. Το ερώτημα το οποίο τίθεται και το οποίο όλοι πρέπει να θέσουμε είναι αναγκαίες και σοβαρές αυτές οι αυξήσεις όταν εμείς ζητάμε από τους λαούς να κάνουν προσπάθειες και θυσίες. Εμείς πρέπει να είμαστε υποδειγματικοί στη διαχείριση του χρήματος και πολύ φοβάμαι ότι το 2016 το παράδειγμα που δίνουμε δεν είναι το σωστό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους, Ινδρικ Ταραντ, για ένα, στο πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ντεπρέ για το ότι συνέταξε με αρκετά μεγάλη συνεργασία με τους συναδέλφους ε, την πρόταση αυτή. Σαν γενναίος ε, καπετάνιος κατάφερε να περάσει το πλοίο της έκθεσης μεταξύ Σκύλας και Χάριβδης. Ε, παρουσιάζω λοιπόν τους, ε, τον κύριο Βέλε και τον κύριο Βίλαντ με αυτά τα αρχαία τέρατα. Οπότε, τρία πράγματα από τους ε, πράσινους. Εμείς θεωρούμε πως τα κτίρια πρέπει να χρηματοδοτηθούν με δανεισμό. Έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια στην ιστορία του ευρώ. Δεύτερον, η αύξηση του επιδόματος γραμματεία ε, μα μοιάζει άκερη και άτοπη αυτή τη στιγμή. Τρίτον, η αύξηση στις δαπάνες πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας φέτος ε, φτάνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Ε, Ήδη όλοι οι βουλευτές ε, αγόρασαν ένα iPad. Ήδη έχουμε, δίνουμε πολλά λεφτά στον κύριο Gates της Microsoft τώρα και στην Apple. Εγώ προτείνω να περάσουμε σε ε, software ανοιχτό, το οποίο είναι δωρεάν και βεβαίως το θέμα εδώ πέρα είναι, ε, είναι σημαντικό. Μιλάω για τα λεφτά. Τέλος και σημαντικό και εγώ θεωρώ πως η μεγαλύτερη απειλή εδώ πέρα είναι η χαμηλά αμοιβόμενη βοηθή παρά κάποιοι ανώνυμοι τρομοκράτες. Οπότε προτιμάω να πληρώνω καλύτερα τους ε, βοηθούς. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σημαντικά τα χρήματα, αλλά και ο χρόνος είναι χρήμα. Λοιπόν, για την, ελευθερία, για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, Μάρκο Βαλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα πλαίσια αυτής της έκθεσης και να το διαβάσετε προσεκτικά λέγεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι υποδειγματικό για να μην απομακρύνεται από την πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν διαρωτώμεθα εμείς γιατί αυξάνονται οι μισθοί των ε, βουλευτών, γιατί αυξάνονται οι δαπάνες των ταξιδιών 3 ε, εκατομμύρια ευρώ επιπλέον και χρειαζόμαστε 15 εκατομμύρια για τους ε, μισθούς ε, των υπαλλήλων που έτσι και αλλιώς πληρώνονται πολύ καλά. Ποιος είναι επίσης ο λόγος για να αυξήσουμε κατά 3,7 εκατομμύρια να αγοράσουμε καινούργια έπιπλα. Νομίζω ότι και η χρηματοδότηση προς τα ιδρύματα τα πολιτικά θα αυξηθεί. Αυτό είναι το παράδειγμα που θέλουμε να δώσουμε στους πολίτες. Αύριο θα δούμε ε, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα κατηγορηθούν γιατί αυξάνουμε το κόστος της λειτουργίας μας. Ευχαριστώ κύριε Βάλια. Ευχαριστώ. Κέλμερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεμπρέ. Τονίστηκε πολλές φορές αλλά εγώ θέλω να το ξαναπώ. Ζούμε σε καιρούς δύσκολους. Τα 550 εκατομμύρια κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν καθημερινά το μήνυμα πως πρέπει να γίνουν οικονομίες. Και μετά θα πρέπει βεβαίως να παίζει και ρόλο υποδειγματικό ο δικός μας ο προϋπολογισμός. Θεωρώ πως θα μπορούσε να περιοριστεί η αύξηση των δαπανών κατά 1,6% και ταυτόχρονα βεβαίως θα πρέπει και να πάμε και πιο χαμηλά από αυτό. Πρέπει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες, ειδικά στον τομέα της πληροφορικής που πρέπει πραγματικά να ε, είμαστε υποδειγματικοί, αλλιώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην έχουμε προβλήματα εδώ πέρα. Από την άλλη είπαμε πως πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την ασφάλεια των κτηρίων. Μην έχουμε όμως ένα φαινόμενο πλασέμπο, δηλαδή να βλέπουμε πράγματα τα οποία μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά, αλλά δεν ενισχύουν την ασφάλεια. Σα ευχαριστώ. Για ένα λεπτό επίση, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Η Ευρώπη έχει πρόβλημα αξιοπιστίας και απόστασης από τους πολίτες. Το λέμε εδώ και χρόνια, είναι μια ανάλυση την οποία επαναλαμβάνουμε και όμως δεν μαθαίνουμε τίποτα. 20 χρόνια το ελεγκτικό συνέδριο απορρίπτει τον ε, προπολογισμό και εξακολουθεί το κοινοβούλιο να τον εγκρίνει. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει τον προπολογισμό της, ενώ τα κράτη-μέλη έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και τώρα μάλιστα ζητάμε να αυξηθεί κατά 1.500 ευρώ το μήνα ο προϋπολογισμός ε, των βοηθών του κάθε βουλευτή. Έτσι δεν θα ενισχυθεί ποτέ ο, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το NVA είναι κατά και θα ψηφίσει κατά και οι υπόλοιποι Φλαμανδοί βουλευτές ε, είπαν ε, το ίδιο, αλλά φοβάμαι πως δεν αρκεί. Αύριο στην ψηφοφορία θα δούμε τι θα κάνουμε για να στείλουμε ένα μήνυμα μεγαλύτερη ευθύνη της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία και HDI. Για ένα λεπτό ο καθένας. Έχω τρεις ομιλητές. Βίκτορ Νεγκρέσκου πρώτος. Για Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πάρω το λόγο ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών διότι έχω απογοητευτεί από την τελική μορφή του κειμένου αν και ο κύριος Δεπρές είναι από τους αγαπημένους μου βουλευτάς. Επειδή όμως εκπροσωπούμε τους πολίτες και δεν θέλουμε τη γραφειοκρατία θεωρούμε ότι δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο κείμενο το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο εφαρμόζει μισθούς ε, βοηθών που είναι χαμηλότεροι για μερικές χώρες μέλη από ό,τι για άλλες. Στην χώρα μου είναι 700 ευρώ μισθός αυτός. Θα ήθελα λοιπόν ίσως να μην μεταφραστεί αυτό που θα πω σε όλες τις γλώσσες γραπτό για να μειωθεί το κόστος, αλλά θέλω να τεθεί το ερώτημα. Η δημοκρατία κοστίζει χρήματα, δεν πρέπει να μειώσουμε τη δημοκρατία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Νότς Μαριές, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θίξω τρία ζητήματα. Πρώτα απ' όλα προβλέπεται από τον προϋπολογισμό μια γραμματιακή ενίσχυση σε ορισμένες επιτροπές. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει καμία ενίσχυση για τη γραμματεία της επιτροπής αναφορών. θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή είναι μια σημαντικότατη επιτροπή η οποία έχει άμεση επαφή και σχέση με τους πολίτες της ευρωπαϊκής ένωσης δέχεται τα αιτήματά τους δέχεται τις αναφορές και είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο άμεσα συνδέεται με τους ίδιους πολίτες. επομένως πρέπει να υπάρξει αύξηση της γραμματιακής ενίσχυσης της επιτροπής αναφορών δεύτερο με προβληματίζει η αντίληψη η οποία λέει ότι πρέπει να περιορίσουμε τον αριθμό των γραπτών ερωτήσεων. βασική δραστηριότητα ενός κοινοβουλίου είναι η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου. εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις τότε είναι προφανές ότι περιορίζουμε τις ίδιες τις αρμοδιότητες που έχουμε θεωρώ λοιπόν ότι είναι υποκρισία να λέμε για δίθεν λόγους οικονομίας ότι πρέπει να μην έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε πολλές γραπτές ερωτήσεις. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Τελευταίος κύριος να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεπρέ για την προσπάθεια που έκανε και να τονίσω αυτό το οποίο ήδη ε, υπόθηκε ότι πρέπει δηλαδή να επενδύσουμε στην ασφάλεια των κτηρίων στις Βρυξέλλες ε, και βεβαίως σε αυτό εδώ πέρα το κτήριο οπωσδήποτε. Αναμφισβήτητο αυτό γιατί είμαστε ένας εξαιρετικός στόχος. Να συμπληρώσω το εξής. Το θέμα της γραμματιακής στήριξης και το θέμα των γραφείων των βουλευτών είναι θέματα τα οποία έχουν προκαλέσει κάποιες συζητήσεις και στη δική μου χώρα και χρειαστήκε να απαντήσω και σε ορισμένα σχόλια τα οποία έγιναν. Είναι ένα θέμα αρκετά ευαίσθητο το οποίο προκαλεί ενδιαφέρον και προς το παρόν αρνητικές αντιδράσεις. Ja, vielen Dank. Ε, Ευχαριστώ κύριε Γιάκοβτσιτς για δύο λεπτά Ζιράρ Ντεπρέ για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω σε δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις που έγιναν. Η πρώτη αφορά τον αριθμό των ερωτήσεων. Μπορούμε πάντα κύριε Μαριά να θέτουμε ερωτήσεις. Δεν τις καταργούμε εντελώς. Απλά περιορίζονται σε πέντε το μήνα αναβουλευτή. 60 δηλαδή μέσα σε ένα κοινοβουλευτικό χρόνο. Το 80% ε, των βουλευτών θέτουν λιγότερες από 60 ερωτήσεις το μήνα και μόνο λιγότερο από 20% θέτουν πάνω του 50% των ερωτήσεων οι οποίες ε, πολλές φορές δεν παρουσιάζουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους πολίτες βέβαια. Κοιτάξτε, εγώ, εγώ έχω το δικαίωμα να λέω την άποψή μου. Αν θέλετε πάρτε μια μπλε κάρτα και να μου θέσετε μια ερώτηση. Τώρα λοιπόν, σχετικά με την εφαρμογή σχετικά με την εφαρμογή της ε, μεταρρύθμισης και μιας καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στους πιστοποιημένους από τη μία συνεργάτες ε, και τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες προβλέπεται η μεταρρύθμιση αυτή να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2016 θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος πιθανώς για έξι μήνες γιατί κάποιοι βουλευτές έχουν υπογράψει συμβάσεις και δεν μπορούμε μονομερός να τις διακόψουμε. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι ε, αν είχα γράψει εγώ το σχέδιο προϋπολογισμού θα το είχα κάνει διαφορετικό. Εγώ βέβαια προσπαθώ σαν εισηγητής για το συγκεκριμένο θέμα να πετύχω μία συνένεση και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στο Προεδρείο. Αυτό σημαίνει συμβιβασμούς. Συμβιβασμός τι σημαίνει. Κάτι το οποίο μου αρέσει και κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Σας ευχαριστώ και για τις κριτικές σας. Ε, είναι πολύ σωστό να έχει κανείς διαφορετικές αντιλήψεις. Αλλά δεν μου αρέσει ο λαϊκισμός και κάποιες παρεμβάσεις αφήνουν να εννοηθεί ότι στον προϋπολογισμό τον οποίο αποφασίσαμε και θα προτείνουμε αύριο για ψηφοφορία πήραμε κάποια μέτρα έτσι ώστε να βάλουν στην τσέπη τους περισσότερα λεφτά οι βουλευτές. Αυτό είναι ψευδές, είναι λάθος και είναι απαράδεκτο. Απλά προσπαθούμε να κάνουμε την εργασία μας με πιο υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο. Η κριτική λοιπόν όταν είναι πολιτικάντικη και λαϊκιστική ε, δεν με συγκινεί. Θα ήθελα να πω ότι διαπιστώνουμε από ορισμένου πολίτες ε, μία απόρριψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλά από αυτά που ακούγονται εδώ τροφοδοτούν αυτή τη στάση. Ευχαριστώ κύριε Ντεπρέ. Τελείωσε η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο.